Καλημέρα σας. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε, λέει η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους. Ε, σήμερα το πρωί θα εξετάσουμε τους διορισμούς και θα ασχοληθούμε με την επιλογή των υποψηφίων για την Προεδρία και τους ανεξάρτητους επίσης, τα ανεξάρτητα μέλη της Εποπτικής Επιτροπής των Κεντρικών Συμβαλωμένων. Ε, προτείνει καταρχήν η, ε, η ίδια η ΕΚΑ η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και στη συνέχεια εμείς αποφασίζουμε. Πρόκειται για τον κύριο Λέμπερ που μας προτείνουν από έναν κατάλογο επικρατέστερων και μετά από τον αύριο του 2019 και μετά από όλη τη διαδικασία επιλογής. Τώρα λοιπόν έχουμε την ανταλλαγή απόψεων με τον ε, επιλεγμένο για την θέση της Προεδρίας βάσει του άρθρου 24α5 του κανονισμού ΕΜΙΡ που ορίζει ότι πριν από τον ορισμό του Προέδρου και των ανεξάρτητων μελών της Εποπτικής Επιτροπής των Κεντρικών Αντισυμβαλωμένων και το πολύ ένα μήνα μετά την επιλογή του Συμβουλίου Εποπτών, ε, το οποίο οφείλει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάλογο με τους επικρατέστερους υποψηφίους ε, που επέλεξε, σεβόμενο την ισορροπία μεταξύ φύλων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από ακρόαση με τους υποψηφίους θα εγκρίνει ή θα απορρίψει την υποψηφιότητά τους. Θα ακούσουμε πέντε λεπτά στην αρχή τον κύριο Λέμπερ και στη συνέχεια θα έχουμε μετά από αυτά τα πέντε λεπτά του κυρίου Λέμπερ θα ακούσουμε τέσσερα λεπτά, ένα λεπτό ερώτηση, τρία λεπτά απάντηση από τον κάθε Ευρωβουλευτή και κάθε πολιτική ομάδα μπορεί να υποβάλει μία ερώτηση. Αν έχουμε χρόνο, στη διαδικασία Catch the θα ακούσουμε περισσότερες ερωτήσεις σύμφωνα με τη στάθμιση και το ειδικό βάρος των πολιτικών ομάδων. Ε, θα ζητήσω λοιπόν από τον κύριο Λέμπερ να ε, μας κάνει στο τέλος μετά από όλα αυτά δύο λεπτά μια μικρή παρέμβαση για να κλείσει. Έχουμε σε 8 γλώσσες διερμηνία σήμερα και για τους διερμηνείς καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να σας μεταφράζουν όταν είσαστε από απόσταση. Γι' αυτό παρακαλώ, λέει Πρόεδρος, να φροντίσετε να μας βοηθήσετε με καλή συνδύση κλπ. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Λέμπερ για τα πέντε λεπτά που έχει για τις αγωγικές του παρατηρήσεις. Έχετε το λόγο κύριε Λέμπερ. Κύριε Λέμπερ, παρακαλώ πατήστε το κουμπί ομιλία. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, είναι τιμή για μένα και προνόμιο βέβαια που βρίσκομαι εδώ σε αυτή την ακρόαση και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Θα μιλήσω αγγλικά. Δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες μάλιστα, έχω εργαστεί στα αγγλικά. Καταλαβαίνω όμως τα γλωσσικά ζητήματα, γι' αυτό και σας λέω καλημέρα σε διάφορες γλώσσες και είπε καλημέρα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά ο κύριος Λέμπερ. Έχω 25 χρόνια που ασχολούμαι με τις χρηματοοικονομικές αγορές και με θέματα κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Και έχω μοναδική εμπειρία στο θέμα αυτό, γιατί έχω ασχοληθεί με τα θέματα αυτά πολύ καιρό από πλευράς εποπτείας και έχω δουλέψει και στο αναλυτικό σκέλος. Γι' αυτό λέω ότι θεωρώ ότι έχω εμπλακεί αρκετά στο ζήτημα. Ξέρω επίσης τις χρηματοπιστωτικές αγορές καλά και έτσι πιστεύω ότι μπορώ να αντιμετωπίσω το θέμα της εποπτείας έξι συστημικών οργανισμών και 60 υποδομών σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Εγώ ίδιος έχω ασχοληθεί με τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους, με διάφορα γραφεία συμψηφισμού και θέλω να τονίσω ότι η εμπειρία που έχω από την εποπτεία και τον έλεγχο είναι κάτι που έχει αναπτυχθεί πολύ και έχουμε καταλήξει σε προδιαγραφές που γίνονται αποδεκτές γενικά. Πριν ήμουνα στο σώμα που κανόνιζε τις προδιαγραφές στη Βασιλεία και έχω ασχοληθεί με τις γενικές προδιαγραφές για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους και έχω ασχοληθεί με θέματα όπως είναι η ανάκαμψη, η εξυγίανση και η αντίσταση των ε, οργάνων αυτών σε πτώχευση. Πιστεύω ότι η γνώση μου από τις χρηματοπιστωτικές αγορές είναι κάτι σημαντικό. Είναι αλήθεια ότι προκύπτουν νέα στοιχεία το θέμα της επάρκειας, της εποπτείας των κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Βλέπουμε όμως ότι έχουμε και θέματα να αντιμετωπίσουμε εξαιτία του Brexit, της διατλαντικής συνεργασίας και υπάρχει βέβαια και η πανδημία. Όλα αυτά είναι προκλήσεις που απαιτούν να προσέξουμε πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι επιπτώσεις στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Έχω πραγματογνωμοσύνη για αυτά τα ζητήματα, όχι μόνο εξαιτία τη συμμετοχή μου στο παρελθόν σε αντίστοιχε θέσεις, αλλά επειδή γνωρίζω καλά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τι ευρωπαϊκέ διαδικασίες και τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δρά για να ενισχύσει την αντοχή των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών. Και επειδή ακριβώς έχω αναμειχθεί σε περίπλοκα ζητήματα, σε διεθνές επίπεδο, ε, πιστεύω ότι είμαι κατάλληλος για αυτή τη θέση. Έχω ασχοληθεί με συνεργετικές δομές, σε επιτροπές, ε, με ρόλο και προέδρου, οπότε προσβλέπω την εμπειρία μου αυτή να τη χρησιμοποιήσω και τώρα στην ε, εποπτική αυτή επιτροπή κεντρικών αντισυμβαλόμενων. Δύο ακόμα στοιχεία θέλω να σας αναφέρω. Πρώτον, Ελπίζω ότι θα μπορέσω να χρησιμοποιήσω τη συνεργατική μου αυτή στάση και από την ηγετική θέση που εφόσον μου επιτρέψετε θα αναλάβω και έτσι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τέλος. Έχω εργαστεί πραγματικά σε διάφορους τομείς με μεγάλη ποικιλομορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχω ηγηθεί ομάδων τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διάφορα στοιχεία και σε διάφορους τομείς. Οπότε ελπίζω η πρόταση αυτή της ε, Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών ε, θα έχει συνέχεια από εσά και έτσι θα μπορέσω να αναλάβω τα καθήκοντά μου χρησιμοποιώντας την προσέγγιση που σας είπα, που είναι ότι θα χρησιμοποιήσω την εμπειρία μου από τους διάφορους τομείς τους οποίους έχω εργαστεί μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα τις ε, ερωτήσεις και απαντήσεις. Ξεκινάμε με την κυρία Ντανούτα Χούμπνερ από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Λέμπερ. Η ερώτησή μου σχετίζεται με αυτά που είπατε. Γιατί εδώ στο Συμβουλίο Εποπτείας έχουμε μία κατάσταση, μια κατάσταση με, μια, με τη δημιουργία μιας νέας δομής σε δύσκολες εποχές. Και εσείς αναφέρατε όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτή την εποχή ως δύσκολη, προβληματική και επιπλέον ε, οι CCP δραστηριοποιούνται παγκοσμίω, οπότε αυτή είναι μια επιπλέον διάσταση που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Εσείς λοιπόν θα βρίσκεστε σε ένα όργανο το οποίο θα δοκιμαστεί σε δύσκολες εποχές και έχετε ήδη κάποια εμπειρία. Έχουν υπάρξει και αναφορές ε, για τις επιδόσεις της CCP κατά τους πρώτους μήνες αυτής της κρίσης και μπορούμε να δούμε σαφώς ότι πέραν ε, της αύξησης των ε, περιθύρων κερδών των παραγόγων έχει παραμείνει ανθεκτική η CCP. Και βάσει του ΕΜΗΡ έχουμε και νέο κανονισμό τώρα και η ερώτηση μου προς εσάς είναι ποιος είναι ο, πώς βλέπετε το ρόλο του Συμβουλίου Εποπτείας ε, τη δομή που είναι εντός της δομής της ΕΣΜΑ Πώς θεωρείτε ότι θα κάνει πιο ανθεκτική, θα γίνει πιο ανθεκτική η CCP ούτως ώστε να μειωθεί η αβεβαιότητα δεδομένου ότι θα υπάρχουν και ε, παραγόντες που θα ε, παρεμποδίσουν τη λειτουργία των CCP. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετική ερώτηση και σας ευχαριστώ. Έχετε δίκιο, είναι δύσκολες εποχές αλλά έχουμε συνηθίσει πια εδώ και καιρό τις δύσκολες εποχές πρέπει να πω. Δεν είναι ακριβώς ε, ό,τι επιθυμούσαμε, αλλά κάτι που βιώνουμε μετά από την τελευταία οικονομική κρίση. Βασικός στόχος ε, του νέου καθεστώτος είναι να βασιστεί σε παρελθούσα εμπειρία, αλλά και να προσπαθήσει να βελτιώσει το σημερινό πλαίσιο, παρέχοντας ένα πλαίσιο περαιτέρω βελτίωσης τη ασφάλεια και τη αποτελεσματικότητα των CCP το πράττει αυτό με διάφορα στοιχεία τα οποία πιστεύω θα αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα και στο σημερινό περιβάλλον το οποίο μας δοκιμάζει γιατί οι νέες δομές πρώτα απ' όλα ενισχύουν την Προεδρία και την, την κοινή χρήση και την διαθεσιμότητα των πληροφοριών, την αλληλεπίδραση και τη σύγκληση των προσεγγίσεων εντός ε, των δομών αυτών όσον αφορά τη CCP. Είναι βασικό να υπάρχει συνοχή στην προσέγγισή μας όταν εξετάζουμε ελλείψει ή ζητήματα που θα μπορούσαν να βελτιωθούν όσον αφορά την ανθεκτικότητα των επιμέρους CCP. Ταυτόχρονα, το νέο πλαίσιο παρέχει επίση επιπλέον εργαλεία όσον αφορά την πιθανή εμπλοκή CCP τρίτων χωρών. Κάτι επίση εξαιρετικά χρήσιμο βάσει παρελθούσα εμπειρία Να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας ε, για την εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο όταν εξετάζουμε κινδύνους που μπορεί να θέσουν στις των χωρών αλλά και για την ε, βελτίωση των ροών πληροφοριών ε, περισσότερο από παλιότερα. Αναφέρατε μια πτυχή των COVID και πολύ σωστά είπατε ότι έχουμε παρατηρήσει να υπάρχουν κάποια προβλήματα και χαίρομαι πρέπει να πω που Συνολικά οι CCP έχουν αποδείξει ότι είναι σταθερή και ανθεκτική, ακόμη και σε τόσο δύσκολες, αβέβαιες ε, και εποχές ε, όπως ζήσαμε στην αρχή της κρίσης του COVID. Ωστόσο πρέπει να εξετάσουμε στενά τις πραγματικές εμπειρίες και υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί, αναφέρατε τα περιθώρια, κάποια ζητήματα που αφορούν τη ρευστότητα, και καλό θα ήταν να ξαναεξετάσουμε περισσότερο τι πιθανέ ε, προκυκλικέ ε, συνέπειε των υπαρχόντων καθεστώτων και υπάρχει και άλλη μια πτυχή που πρέπει να αναφερθεί αυτό που ζήσαμε ε, όσον αφορά τι αντιδράσεις για τον COVID τα σενάρια εργασίας από το σπίτι όσον αφορά ορισμένα CCP διότι δημιουργούν νέα ευάλωτα σημεία για κυβερνοεπιθέσεις όλα αυτά απαιτούν καλή ανάλυση και απόκριση αναγκαία ώστε να, ρυθμιστεί, να ρυθμιστούν λεπτομέρειε τη μία ή τη άλλη πτυχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα έχουμε την Evelyn Regner από τους σοσιαλιστές. Ε, Miss Regner will uh, take the floor a bit later, so you can go to the next. Κυρία Ρέγνερ μπορεί να πάρει το λόγο, οπότε περνάμε στον επόμενο μιλητή. Οπότε, η Μόνικα Σεμέντο τώρα από το Ρινιού έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Λεμπέ. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας σήμερα. Η ερώτησή μου είναι... Views between the ECB. Καταρχήν να πω ότι στο παρελθόν υπήρχε μια διαφορά απόψεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, και ΕΣΜΑ σε ό,τι αφορά τα equivalence regimes. Σε ό,τι αφορά λοιπόν και την αβεβαιότητα που ισχύει, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας μελλοντικά με το Ηνωμένο ε, Βασίλειο, ε, πώ θεωρείτε εσείς πω θα πρέπει να λαμβάνει η χώρα η αντιμετώπιση των εθνικών CCP έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε και τη δημοσιονομική και οικονομική σταθερότητα. Δεύτερον, πείτε μας εσείς βάσει την εμπειρία που έχετε ε, σε επίπεδο εποπτείας πώς θα μπορούσε ο εποπτικός ακριβώς τομέας να συμβάλλει ε, και επίσης πώς εσείς από την πλευρά σας θα προωθήσετε ε, την ισόρροπη εκπροσώπηση των φίλων στην ΕΣΜΑ και από εκεί και μετά ποιες σημαντικές αλλαγές θα θέλατε να λάβουν χώρα στην ίδια την ΕΣΜΑ έτσι ώστε να βελτιωθεί το gender balance, η ισόρροπη δηλαδή εκπροσώπηση των φίλων εκεί. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Λόβε. Ε, είναι αρκετά περίπλοκο το ερώτημα και η απάντηση δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τη δώσω σε 3-4 λεπτά, αλλά να προσπαθήσω. Πράγματι αυτό που είπατε ε, ως προς την ε, σχετικά πρωτόγνωρη κατάσταση την οποία έχουμε να κάνουμε, δηλαδή ένα μεγάλο οικονομικό κέντρο εκτός πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στο εγγύς μέλλον εκτός ε, και της ε, νομοθετικής αν θέλετε αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει ε, και θα πρέπει να το εξετάσουμε από πλευράς οικονομικής σταθερότητας. Νομίζω πως το νέο πλαίσιο ΕΜΙΡ δημιουργεί ακριβώς ένα καλό σημείο αφετηρία σε ό,τι αφορά πάντοτε την πτυχή της οικονομικής σταθερότητας, έτσι ώστε δηλαδή να διασφαλίσουμε ότι δυνητικές επιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον κατάλληλο τρόπο. Ωστόσο, εδώ τώρα έχουμε μία έκτακτη περίπτωση. Δηλαδή, μία περίπτωση όπου μπορεί να υπάρξουν πολύ βίαιες αλλαγές, ακριβώς επειδή βλέπουμε να βρισκόμαστε κοντά στην εκπνοή της ε, ε, προθεσμίας ε, για την επίτευξη μιας συμφωνίας. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι άμεσες επιπτώσεις και τι ακριβώς θα χρειάζεται σε ό,τι αφορά ε, τα ε, κράτη-μέλη για την πρόσβαση σε διεθνείς ε, αγορές και προκειμένου να αποφύγουμε τον καταγερματισμό σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα. Βρισκόμαστε σε φάση ακριβώς τώρα δοκιμαστική προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα σύστημα με πολύ μικρές καθυστερήσεις. Πέραν όμως αυτών των βραχυπρόθεσμων λύσεων θα πρέπει να δούμε και ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να επιτύχουμε την εξορρόπηση δύο διαφορετικών πτυχών. Η μία από αυτές είναι η δυνατότητα για τους ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν τη δυνατότητα να πρόσβαση στις ε, παγκόσμιες αγορές και από την άλλη πλευρά υπάρχει και ε, το, το νόμο αν θέλετε συμφέρον της κυριαρχίας οπότε εδώ τίθεται το ερώτημα και, το, και θα πρέπει δηλαδή να δούμε το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει πιο άμεσα τέτοιου είδους ε, ε, διαδικασίες. Και βέβαια εδώ θα χρειαστεί να υπάρξει και μια κανονιστική, αν θέλετε, ευθυγράμμιση καλύτερη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Σε κάθε περίπτωση αυτό που χρειάζεται είναι μια ξεκάθαρη ανάλυση των επιπτώσεων σε ό,τι αφορά την οικονομική σταθερότητα και σε σχέση, για παράδειγμα, με το relocation και το non-relocation και αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πολιτική συγκεκριμένη και την οποία μάλιστα θα ανακοινώσουμε και θα κοινοποιήσουμε σε όλους με τον κατάλληλο τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε δηλαδή να επιτύχουμε την κατάλληλη προετοιμασία των ε, αγορών και των σχετικών υποδομών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δική μου εμπειρία, όπως ε, γνωρίζετε αυτή η εποπτική οι εποπτικές αρμοδιότητες ε, εδώ στην ΕΣΜΑ είναι συμπληρωματικέ ε, ε, προς αυτό το θέμα και εγώ έχω γνωμοσύνη σε ό,τι αφορά την εξέταση της ασφάλειας και την αποτελεσματικότητα των κεντρικών αντισυμβαλόμενων τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και πέρα αυτής. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το Margin Collateral Settlement, Interoperability και τέτοιου είδους στοιχεία είναι αυτά που μας έχουν απασχολήσει ό,τι αφορά τις ε, κεντρικές τράπεζες. Και βέβαια ακριβώς ε, λόγω και της εμπειρίας ε, που έχω στον τομέα της, των δραστηριοτήτων της Κεντρικής Τράπεζας έχω αυτή την εμπειρία σε ό,τι αφορά τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους. Σε ό,τι αφορά τώρα το τελευταίο ερώτημα που θέσατε, θεωρώ πως πραγματικά η διαφορετικότητα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο μπορεί να εμπλουτίσει και να ενισχύσει ε, την λειτουργία οποιοδήποτε οργανισμού. Και εδώ αναφέρομαι λοιπόν στην διαφορετικότητα όχι μόνο σε ό,τι αφορά το φύλλο, αλλά σε, ε, από κάθε διάσταση. Και σε όλη μου τον επαγγελματικό ε, βίο, οι ομάδε στον οποίο εγώ ηγούμε, πάντοτε πράγματι απηχούν αυτή την ανάγκη εξ ισορροπημένης εκπροσώπησης όλων των διαφορετικών πτυχών, δηλαδή φύλου, εθνότητας, υπηκότητας και ούτω καθεξής. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω πως με αυτή τη διαφορετικότητα υπάρχει αύξηση της παραγωγικότητας και είναι καλύτερη λήψη των αποφάσεων. Και αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο της δικής μου ιεραρχίας ε, ε, τα δύο τρίτα ε, είναι γυναίκες και το 70% των εφεσταμένων είναι επίσης γυναίκες. Οπότε νομίζω εδώ έχουμε πλέον ένα ζήτημα εξορρόπησης από την ανάποδη. Επίσης επιτρέψτε μου να πω ότι η ΕΣΜΑ πράγματι έχει λάβει σοβαρά υπόψη της την ανάγκη του να υπάρχει ισόρροπη εξορρόπηση των δύο φύλων. και πράγματι η, η, τα κεντρικά διοικητικά στελέχη του Υποπτικού Συμβουλίου έχουν πάντοτε κατά νου αυτή την ε, πτυχή. Και αναμένω βέβαια εδώ με μεγάλο ενδιαφέρον τη συνεργασία με τους συναδέλφους, καθώς ε, θεωρώ πως ε, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την διαφορετικότητα εντός της ΕΣΜΑ. Ευχαριστούμε πολύ να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε περιορισμένο χρόνο. Ήδη έχουμε κάποια μικρή καθυστέρηση, οπότε αν θέλουμε να τηρήσουμε το χρόνο μας πρέπει να προσέχουμε. Τώρα η ομάδα ID δεν μου έχει δώσει όνομα. Αν υπάρχει κάποιος που θέλει να πάρει το λόγο, ευχαρίστως από το ID. Αλλιώς Σβέν Γκίγκορτ είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κύριε Λούμπερτ. Ελπίζω να με ακούτε καλά. Έχω μία κυρίως ερώτηση. Αν δείτε πόσο τεχνικό είναι το ζήτημα, το οποίο βέβαια εσείς γνωρίζετε καλά, είσαστε εξοικειωμένος, υπάρχει ο ρυθμιστικός κίνδυνος. Το είδαμε αυτό και στο αδερφό ε, όργανο με σας. Και υπάρχει εδώ πέρα ζήτημα σχεδιασμού. Οπότε ρωτάω, τι μέτρα εσείς θα πάρετε για να αποφύγετε αυτό το regulatory capture, ιδιαίτερα μετά από τις πρόσφαστες ε, συστάσεις της Ombudswoman για την περίπτωση του κύριου Φάρκας Πώς θα διασφαλίσετε δηλαδή, δεδομένου ότι είναι τόσο τεχνικό το ζήτημα, πόσο θα διατηρείτε απόσταση από εκείνους για τους οποίους θα είσαστε εσείς υπεύθυνο να ρυθμίζετε. Ευχαριστώ. Κύριε Γκυγόλ, πράγματι αναφέρεστε σε ένα πολύ θεμελιώδες ε, ζήτημα, λέει ο κύριος Λέμπερ. Και όντω πρόκειται για μια κλειστή κοινότητα όταν έχουμε να κάνουμε με συμψηφισμό, με κεντρικούς ε, αντισυμβαλόμενου και με την τεχνικότητα του ζητήματος. Όντως, εδώ θα πρέπει κανείς να ξεχωρίσει τις καθαρά τεχνικέ ε, πτυχές ε, που έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση και την ανάλυση και που εννοείται απαιτούν υψηλή ικανότητα από πλευράς της ΕΣΜΑ, της Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, ώστε να λαμβάνει υπόψη όλες τις πτυχές που έχουν να κάνουν με τους κινδύνους. Και αυτό είναι κάτι που προσέχω όλος ιδιαίτερος. Συγχρόνως όμως, πρέπει να υπάρχει και διάλογος με τις εποπτικές αρχές για να δούμε τι είναι αυτό που βοηθάει στη νέα δομή. Πρώτα απ' όλα βοηθάει η λογοδοσία, η αλληλοεπίδραση πέρα από την ίδια την ΕΣΠΑ, δηλαδή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ θα το φροντίσω αυτό. Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι να μην ξεχνάμε τη διάσταση της πολιτικής. Και εδώ θα φροντίσω να χρησιμοποιήσω την εμπειρία που έχω συλλέξει μέχρι τώρα και σε θέματα πολιτικής και έτσι να μπορώ να εξετάζω τα θέματα από πλευράς σταθερότητας Στο παρελθόν ήμουν τυχερός γιατί μπόρεσα να ελέγξω διάφορους τομείς υποδομών και για παράδειγμα τα συστήματα πληρωμών που είναι κάτι περισσότερο του δημόσιου. Οπότε αυτό το οποίο είναι εδώ κλειδί είναι να διατηρήσουμε την αναγκαία απόσταση, συγχρόνως όμως να υπάρχει διαφάνεια Και αυτό το κάνω και φαίνεται και από το παρελθόν μου και από το πλαίσιο το οποίο υπάρχει στην ΕΣΜΑ σήμερα, ώστε να υπάρχει αρκετή διαφάνεια για τις αλληλοεπιδράσεις και να είμαστε και ανοιχτοί απέναντι στις διάφορες πλευρές και από πλευράς των κεντρικών αντισυμβαλόμενων και των ε, οντοτήτων που εκαθαρίζονται, αλλά και με εσά. Διαβεβαιώ ότι θα υπάρχει διαφάνεια στη θητεία μου. Ευχαριστούμε. Γιώχαν Φανόβερφελτ, ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Διάβασα με ενδιαφέρον το βιογραφικό του υποψηφίου και δεν θεωρώ ότι μπορούμε να αμφισβητήσουμε τις ικανότητές του, οπότε θα εστιαστώ σε κάποια γενικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, τι λέτε στους κριτικούς που θεωρούν ότι έχουμε ένα στρατό μόνο με στρατηγούς και όχι στρατιώτες. Ε, τι θα γίνει με το τεχνικό προσωπικό που θα σας βοηθήσει στην εποπτεία των CCP εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η τρίτη ερώτηση, σε τι θα εστιαστείτε αφού ο φόρτος εργασίας περάσει από τη μεταβατική φάση, ληφθούν οι βασικές αποφάσεις και περάσει η εργασία στο κανονική εργασία, όπως το ονομάζουμε, normal business. Ευχαριστώ πολύ. βασικά σημεία και αυτά τα οποία έχω διαρωτηθεί και εγώ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν χρειαζόμαστε μόνο αρχηγούς, χρειαζόμαστε και εμπειρογνώμονες ε, στην πραγματική ζωή. Μία πτυχή Εγώ είμαι καθισχασμένος γιατί το πλαίσιο, το νέο πλαίσιο που έχουμε αναγνωρίζει αυτή την ανάγκη και αναφέρεται στην ανάγκη επαρκούς ε, στελέχωσης. Εγώ λοιπόν θα συζητήσω ενδελεχώς ε, με την ε, ανώτατη διοίκηση της ΕΣΜΑ για το πώς μπορεί να γίνει όλο αυτό και τι απαιτείται, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα καθήκοντα της εποπτικής, του Εποπτικού Συμβουλίου θα μπορέσουν να εκτελεστούν σωστά. Είναι μια κατάσταση που γνωρίζω πολύ καλά και στη σημερινή μου θέση και στις παλιές μου θέσεις την έχω βιώσει. Ε, πρέπει, είναι κάτι που πρέπει να υπερασπίσει διαρκώς και να προβάλλεις διαρκώς, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα καταφέρουμε να παρέχουμε μια καλή και αιτιολογημένη εξήγηση όσον αφορά τις δεξιότητες που απαιτούνται εντός της ομάδας για να υποστηριχθεί η πολυμορφία των καθηκόντων που ε, θα έχει στην αρμοδιότητα της είναι το νέο υπόπτικο συμβούλιο. Υπάρχει μια πτυχή που αναφέρατε. Πρώτα απ' όλα βρισκόμαστε σε εξαιρετικές ε, συνθήκες δεδομένων όλων των δυσκολιών. Πρέπει λοιπόν να οριστούν ε, προτεραιότητες ε, και να εστιάσουμε τις προσπαθίες μας και απαιτούνται ιδιαίτερες προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσκολίες βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα με τον κατάλληλο τρόπο. Τα καθήκοντα τα οποία εκχωρούνται στο Εποπτικό Συμβούλιο είναι τέτοια που είμαι βέβαιος ότι δεν πρόκειται να βαρεθεί κανείς. Με την άμεση σύσταση αυτού του νέου καθεστώτος έχουμε επαρκή μέσα για να ε, πραγματοποιούμε αξιολογήσεις τακτικά, να κάνουμε τα stress test, να υπάρχει και χρόνος να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και να ενισχύσουμε περαιτέρω τη σύγκληση ειδικότερα ε, ε, εντός της ευρωπαϊκής εποπτείας τη εποπτείας των CCP εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, αφού περάσει το πρώτο stress test, ε, δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα γίνει αυτό, θα υπάρξουν ευκαιρίε ώστε να διασφαλιστούμε ότι όλοι θα μπορούν να εργαστούν και θα έχουν αρκετή δουλειά προχωρώντα και προ το μέλλον. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τώρα δίνω το λόγο στην Εβελίν Ρέγνερ από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Εσείς ως πρόεδρος θα συμβάλλετε στην ανάπτυξη του προγράμματος εργασίας της ΕΣΜΑ, στους στόχους και στις προτεραιότητες. Και η ερώτησή μου είναι πώς θα προωθήσετε την προστασία των επενδυτών, την οικονομική σταθερότητα δεδομένης της κλιματικής αλλαγής και της σημερινής ε, κρίσης υγείας που αποτελούν κινδύνους για την παγκοσμία οικονομία και πέραν αυτών ε, σκάνδαλα όπως το Wirecard οδηγούν σε απώλεια εμπιστοσύνη, ειδικότερα των μικρών μετόχων. Δεδομένων αυτών των προκλήσεων, κατά τη δική σας άποψη, ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που απαιτούνται για την ε, χρηματοπιστική σταθερότητα και να διασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν ε, δύο διαφορετικέ ε, πτυχέ σε σχέση με αυτό που ρωτήσατε. Καταρχήν, το ζήτημα τη ε, προστασία των επενδυτών είναι κάτι το ευρύ ω ζήτημα. Και κινείται δηλαδή πέραν τη εστίασή μα στου κεντρικού αντισυμβαλούμενου. Αντιλαμβάνομαι όμω ότι πρόκειται για κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Και από εκεί και μετά βλέπουμε ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε κάποιες ε, θεμελιώδεις μας προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά την εποπτεία για να αντιληφθούμε δηλαδή και το τι ακριβώς ε, πού θα πρέπει να εστιάζουμε σε ό,τι αφορά τις εποπτικές μας δραστηριότητε. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά δηλαδή το εύρος των κανονιστικών παραμέτρων έτσι ώστε να μην υπάρχουν να μην εστιάζουμε σε, σε λανθασμένες ε, λειτουργίες και αντιθέτως να εστιάζουμε σε εκείνες που έχουν πραγματικές επιπτώσεις για τους ε, ε, καταναλωτές. Να αποφύγουμε δηλαδή εποπτικές λειτουργίες οι οποίες τελικά βρίσκονται και εκτός του, της αρμοδιότητας και του πεδίου το οποίο καλύπτουν οι κανονιστικές αρχές. με αυτόν τον τρόπο δηλαδή έχουμε προσπαθήσει να κινηθούμε σε ό,τι αφορά τις εποπτικέ μας δραστηριότητε. Τώρα σε ό,τι αφορά τη δεύτερη πτυχή ε, στην οποία αναφερθήκατε, είναι κάτι το οποίο μας ε, απασχολεί πολύ, δηλαδή η βιωσιμότητα σε ό,τι αφορά την ε, εξέταση και την παρακολούθηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Πέραν δηλαδή και των ε, CCP των κεντρικών αντισυμβαλόμενων θα προσπαθούμε πάντοτε να έχουμε ε, το νου μας γιατί και οι ε, αντισυμβαλόμενοι μπορούν για παράδειγμα και εκείνοι να δεχθούν τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή αλλά από εκεί και μετά ευρύτερα υπάρχει η ανάγκη οι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι οι ίδιοι να αναγνωρίσουν αυτή την κατάσταση και να είναι σε θέση από μόνο τους να αναγνωρίζουν τους κινδύνους οι οποίοι μπορούν να προκύψουν από την κλιματική αλλαγή. Προκειμένου δηλαδή ακριβώς αυτή οι κίνδυνοι να λαμβάνονται υπόψη και στα μοντέλα αξιολόγησης κινδύνων τους. Επίσης θα προσπαθήσουμε σε αυτόν τον άξονα να αναπτύξουμε μια στοχευμένη υπηρεσία, για παράδειγμα δηλαδή σε ό,τι αφορά τα ζητήματα βιωσιμότητας ε, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την προσφορά νέων προϊόντων που βασίζονται ακριβώς σε εργαλεία refinancing αναχρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Δεν βλέπω ε, να υπάρχει κάποιος συνάδελφος από την ΚΟΕ που να έχει δει στο λόγο. Οπότε θα δώσω τον λόγο στον κύριο ε, Λόβε για να κάνει ε, κάποια καταληκτικά σχόλια. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για όλα αυτά τα εξαιρετικά ερωτήματα. Ε, θα αποτελούσε μεγάλη μου χαρά να επιλεγώ σε αυτή την θέση και να συνεχίσω τον διάλογό μας για αυτά τα ζητήματα. Ένα βασικό ζήτημα που τίθεται είναι το ότι η προ κλήσεις οι οποίες αναφέρθηκαν σε αυτά τα ερωτήματα είναι πολυπίκυλες και αφορούν το μέλλον των αγορών συνολικά. Τέτοιου είδους λοιπόν πολυσχεδία ερωτήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω ενός πλήρους ευρέως διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων ε, θεσμικών οργάνων αλλά και φορέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός αυτής. Οπότε εγώ λοιπόν από τη δική μου πλευρά θα ήμουν διατεθειμένος ε, να συμβάλλω ε, και με, την, με τις δικές μου σκέψεις και στο πλαίσιο βέβαια ακριβώς αυτής της θέσης, αν μου δοθεί δηλαδή, του Προέδρου της Αποπτικής αυτής αρχής για τους Κεντρικούς αντισυμβαλόμενους. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα περιμένουμε λίγα λεπτά για να μπορέσουμε να έχουμε τον επόμενο υποψήφιο, την επόμενη υποψήφια και τότε θα ξεκινήσουμε με την επόμενη ακρόαση. Chair, the, the, the candidate, Ms. is connected, so Ωραία. Μπορούμε να περάσουμε στην κυρία Νικολέτα Τζούστο, την επόμενη υποψήφια που προτείνεται για μία από τις δύο θέσεις ανεξάρτητων μελών της νέας Εποπτικής Επιτροπής για Κεντρικούς Αντισυμβαγόμενους. Ε, αποφασίσαμε στις 27 Αυγούστου του 2020 όσον αφορά την απόφαση επιλογής της κυρίας ε, Τζούστο που ενέκρινε με κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων ίδια η ΕΣΜΑ εφόσον ε, δημοσιεύτηκαν οι κενές θέσεις τον Νοέμβριο του 2019. Η ανταλλαγή αυτή απόψεων με την επιλεγμένη υποψήφια της Εποπτική Επιτροπής Κεντρικών Συμβαλόμενων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού ΕΜΗΡ και θα γίνει κάτω από τι ίδιε συνθήκε που έγινε και η προηγούμενη ακρόαση. Θα έχουμε δηλαδή μια εισαγωγική παρέμβαση τη κυρία Τζου στο 5 λεπτών και στη συνέχεια θα έχουμε ερωτήσει και απαντήσει. Ένα λεπτό η κάθε ερώτηση και τρία λεπτά για την κάθε απάντηση. Και μετά στο τέλος η υποψήφια θα μπορέσει και πάλι να πάρει το λόγο. Συνεπώς, δίνω το λόγο στην κυρία Νικολέτα Τζούστο τώρα παρακαλώ για τις εισαγωγικέ της παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Όπως είπε και η Πρόεδρος, ονομάζομαι Νικολέτα Τζούστο και είμαι επικεφαλής της υπηρεσίας ε, διεθνών σχέσεων στην Κόντσαπ, που είναι ο Ιταλός ρυθμιστής. Εδώ και χρόνια εργάζομαι σε αυτή τη θέση, όπως βλέπετε προφανώς και από το βιογραφικό μου. Και έχω μεγάλη εμπειρία στο διεθνή χώρο και ιδιαίτερα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ήδη από τις σπουδές μου εργάστηκα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνέχεια ασχολήθηκα με την προσχώρηση της Ρουμανίας, επειδή είμαι από εκεί. Έχω συντάξει και εκθέσεις για ομοτήμους από πλευράς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και έχω συνεργαστεί με διάφορες ομάδες σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, την Ιόσκο, για παράδειγμα σε επίπεδο Ιόσκο. Και έχω πραγματογνωμοσύνη επίσης στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας. Όσον αφορά το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους, δεδομένου ότι για τέσσερα χρόνια ήμουν πρόεδρος της μόνιμης Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών προκάτοχος ουσιαστικά αυτού που δημιουργούμε τώρα ως Εποπτική Επιτροπή για Κεντρικούς Αντισυμβαλόμενους. Και σίγουρα θα ασχοληθούμε και με επιτροπές στα πλαίσια του κανονισμού ΕΜΙΡ. Σίγουρα η εποπτεία και οι αρμόδιες εποπτικές ε, αρχές ε, θα είναι σε επαφή μαζί μας και εμείς μαζί τους. Οπότε, να σας πω επίσης ότι πέρα από αυτό έχω εμπειρία στη διεθνή συνεργασία. Έχω εργαστεί για την ΕΣΜΑ στα πλαίσια του Brexit, έχοντας ετοιμάσει διάφορα μεμοράντα σχετικά με τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους, έχω ασχοληθεί με ανταλλαγή πληροφοριών ε, όσον αφορά το τι θα γίνει μετά το Brexit. Έχω συγκεκριμένη εμπειρία στη διεθνή συνεργασία. γιατί είμαι αρμόδια να επεξεργάζομαι ε, τα αιτήματα που μας φτάνουν και το ίδιο θα χρειαστεί και στα πλαίσια του ΕΜΙΡ. Για ε, κεντρικούς αντισυμβαλόμενους από τρίτες χώρες σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει ε, ανανέωση του μνημονίου κατανόησης που υπάρχει μεταξύ μας και η νομοθεσία του κανονισμού ΕΜΙΡ μιλάει για το δικαίωμα πρόσβασης από τρίτες χώρες και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι συλλεγμένες πληροφορίες. και τα στοιχεία. Σύμφωνα πάντα με τις διαδικασίες που βρίσκονται ενισχύ. Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να εξαντλήσω το χρόνο μου. Νομίζω ότι έχω φτάσει στα πέντε λεφτά. Οπότε πείτε μου αν μπορώ να συνεχίσω ή να σταματήσω και να προχωρήσουμε με ερωτήσεις και απαντήσεις. Τι λέτε. Πρόεδρο, σε ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως, μπορούμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις και στις απαντήσεις. Και ξεκινάμε με την κυρία Ντανούτα Χούμπνερ από το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Όπως αναφέρατε το Brexit, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση για αυτό το θέμα, για το Brexit και για τις αποφάσεις ισοδυναμίας, αντιστοιχίας. Η ερώτησή μου σχετίζεται με το ότι η, το Συμβουλίο Υποπτίας θα έχει και καθήκοντα ρυθμιστικά, εποπτικά για τρίτες χώρες επίσης, για δικαιοδοσίες που έχουν δηλωθεί ως αντίστοιχες. Και ξέρουμε ότι η βασική γραμμή των Βρετανικών αρχών ε, όσον αφορά πολιτικά θέματα και των αρχών που αφορούν τις εκαθαρίσεις ήταν το να επανακτήσουν τον έλεγχο το να αναχωρήσουν ουσιαστικά, να απομακρυνθούν από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Στο πλαίσιο αυτό η ερώτησή μου είναι, έχουμε δύο επιλογές. Πώς ε, βλέπετε εσείς τα υπέρ και τα κατά των δύο επιλογών. Ε, η μία επιλογή είναι εξάντε εκ των προτέρων να τραβήξουμε μια γραμμή πέραν της οποίας ε, μια δικαιοδοσία δεν θα θεωρείται ισοδύναμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον το θεωρείτε εφικτό και τι ωφέλη θεωρείται ότι θα μπορούσε να έχει και τι μειονεκτήματα ενδεχομένως. Και η δεύτερη επιλογή είναι να χορηγήσουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο για συγκεκριμένα ζητήματα μία ισοδυναμία περιορισμένη χρονικά. Η ερώτηση προς εσάς είναι ποια λύση προτιμάτε για να είναι πιο αποτελεσματική η δράση μας, πιο αποδοτική και για να έχουμε και σταθερότητα κάτι που είναι ζητούμενο μέσα σε τέτοιες διαφορετικές προσεγγίσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Είναι πολύ βασική. Βασικό το θέμα ισοδυναμία παραμένει ένα από τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας. βασίζεται στην αναγνώριση των CCP και αποτελεί προϋπόθεση. Τώρα υπό το EMIR 2, ευτυχώς, το σύστημα έχει μεγαλύτερη ευελιξία και υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της ισοδυναμίας που θεωρεί το δεδομένη στο προηγούμενο καθεστώς. Και επίσης υπάρχει και η συγκριτική συμμόρφωση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, διότι αφενός έχουμε τις ισοδυναμίες ρέμπους εξάντυπους ε, την ανάλυση του νομικού καθεστώτος ενώ η συγκριτική συμμόρφωση σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε και τις λεπτομέρειες της συμμόρφωσης ε, ενός συγκεκριμένου CCP με τους κανόνες όπως έχουν σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή προσωπικά δεδομένη της κατάστασης και λαμβάνοντας επίσης υπόψη το ότι όποτε έχεις να κάνεις ε, με σχέσεις με τριτές χώρες πρέπει να λαμβάνεις υπόψη και τα πτυχές ε, τα που τα αντί, τυχόν αντίπεινα ε, και που μπορεί να επηρεάσουν τις συναλλαγές στην Ευρώπη σε εποχές που δυστυχώς εξακολουθούν ε, να μας βρίσκουν όλους σε στενή συνεργασία διότι ξέρουμε όλοι ότι πάντα ζητούνται διάμεσα βήματα πιστεύοντας ότι τελικά θα δοθεί μια θαυματουργή λύση. Εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε αυτή την ισοδυναμία υπό όρους και με χρονικό περιορισμό που θα μας επιτρέπει την απαραίτητη ευελιξία ώστε να διασφαλίζουμε ε, συνθήκες ίσου ανταγωνισμού, επαρκή προστασία των ευρωπαϊκών αγορών και των ευρωπαϊκών φορέων διότι οι δουλειές πρέπει να συνεχίζουν να γίνονται και και ο χρόνος ε, δεν είναι άφθονος. Έχουμε ελάχιστο χρόνο μέχρι τα τέλη του έτους, αλλά ευτυχώς το ΕΜΗΡ έχει ε, προσθέσει κάποιο επίπεδο ευελιξία στο νομοθετικό μας πλαίσιο. Δεν είναι ακόμα όσο ευέλικτο είναι άλλα, ε, άλλες αρμόδιες αρχές όπως οι, οι αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. όπου μπορούν εντό λεπτού να αποφασίσουν να αναλάβουν μια δράση. Εδώ θα υπάρχει έσμα, η επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η επαφή επίσης με το πολιτικό επίπεδο που εκπροσωπείται από εσάς και το Συμβούλιο. Κατά βάση αυτή είναι η πρώτη μου απάντηση και ευχαρίστω να την αναλύσουμε περισσότερο αν το επιθυμείτε. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα Χωνός Φερνάντες από τους Σοσιαλιστές. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ σε αυτή την ακρόαση. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτή, αυτές οι ακροάσεις είναι η απόδειξη ότι ε, μπορούμε να έχουμε εξαιρετικούς ε, υποψηφίους. Ε, θέλω να συγχαρώ, να συγχαρώ λοιπόν την ΕΣΜΑ για τον κατάλογο τελικών υποψηφίων. Ουδέποτε έχουμε δει τόσο καλού υποψηφίου. Σε κάθε περίπτωση, η ερώτησή μου προ εσά έχει ω εξή. Σήμερα η Επιτροπή αυτή θα ψηφίσει βάσει των ε, κριτηρίων που πρέπει να λάβει υπόψη η ΕΣΜΑ για να καθορίσει κατά πόσο η κεντρική αντισυμβολόμενη ε, τρίτων χωρών είναι συστημικά σημαντική ή μπορεί να γίνουν ε, συστημικά σημαντικοί για την χρηματοοικονομική σταθερότητα στην Ένωση. Εγώ ανησυχώ για αυτή την κατάσταση. Η ομάδα μου σε κάθε περίπτωση θα υποστήριξει την πρόταση της Κομισιόν, αλλά έχουμε κάποιες αμφιβολίες για τη χρήση των ε, ποσοτικών κατοφλίων για την ανάλυση των CCP συστηματικά ισχυρότερο, θα έλαμε μια πιο ισχυρή ποιοτική προσέγγιση ούτως ώστε να καθορίζεται κατά πόσο μια e CCP μπορεί να εφαρμόσει του ευρωπαϊκούς κανόνες. Θα ήθελα να μου πείτε, γνωρίζετε ε, τα γνωρίζετε αυτά τα θέματα και θέλω να μου πείτε την άποψή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την ε, ερώτηση αυτή θα θυμάται το Κοινοβούλιο ότι η απάντηση που αρχικά είχε προταθεί από την ΕΣΜΑ ε, ήταν να επιμείνουμε περισσότερο στα ποιοτικά κριτήρια. Βέβαια τα ποιοτικά κριτήρια συνοδεύονται από υψηλότερη διακριτική ευχέρεια και υπήρξε εδώ αντίδραση από τον κλάδο και όχι μόνο από αυτόν και από άλλες δηλαδή από την πλευρά άλλων συναρμόδιων αρχών. Ε, δηλαδή η Ιώσκο, και άλλοι για παράδειγμα σε διεθνέ επίπεδο αντέδρασαν σε σχέση με αυτήν την ε, ε, πρόταση και βέβαια το ζήτημα των διεθνώς αναγνωριζόμενων κεντρικών αντισυμβαλόμενων από την πλευρά των κρατών και βέβαια τίθεται το ζήτημα εδώ γενικότερα του πώς είναι δυνατόν να ε, γίνεται έλεγχος των αποφάσεων που λαμβάνει εδώ εκαστοτε αρμόδια αρχή και σε συγκεκριμένη περίπτωση από την ΕΣΜΑ και σε ορισμένες περιπτώσεις από τις κεντρικές τράπεζες. αφού βέβαια είναι σημαντικό να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζονται και οι κεντρικέ τράπεζε για τέτοια ζητήματα. Εγώ προσωπικά θα προτιμούσα να υπάρχει κάποια μεγαλύτερη ευελιξία. Από την άλλη πλευρά ε, θεωρώ ότι εδώ πρόκειται για μια περίπτωση όπου μαθαίνουμε ε, εφαρμόζοντας ε, τα όσα κάνουμε στην πράξη. Ε, και αυτές οι αντιρρήσεις ε, στις οποίες αναφερθήκατε ίσως ε, να αποτελούν ακριβώς αυτό τον, τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια να υπάρξει περισσότερη ασφάλεια δικαίου σε ό,τι αφορά δηλαδή και τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξωτερικούς εταίρους. Πρόκειται δηλαδή εδώ για ένα σημείο αφετηρίας, κάτι δική μου άποψη και, κάτι, και θεωρώ εγώ ότι ε, η υποχρέωση εδώ που έχουμε και η δυνατότητα που μας δίνουν τα ε, εκτελεστικά μέτρα είναι ότι μπορούν να διορθωθούν. Άρα λοιπόν σε επίπεδο Ευρώπης θα πρέπει να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες ως προς τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε το τι συμβαίνει στον κλάδο, να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις και έτσι ε, να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ποια είναι τελικά η συστημική συνέφεια αυτό το ε, systemic relevance και σε σχέση και με το relocation. Εγώ θεωρώ δηλαδή πως αυτή η διαδικασία θα τρέξει με βάση διαφορετικές φάσεις και θα υπάρξει βέβαια και κατάλληλος, έλεγχο έλεγχος σε πολιτικό επίπεδο. Συχνά δηλαδή εξετάζουμε τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους ως, έναν, ως φορείς οι οποίοι ουσιαστικά ε, δρούν αυτόνομα και θα πρέπει να εξετάζουμε τις ε, δυνατότητες που έχουν να λαμβάνουν αυτόνομα αποφάσεις. Ωστόσο, ε, υπάρχει και η άλλη πτυχή, ότι δηλαδή αυτοί οι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι αποτελούν πολύ σημαντικέ ε, πλατφόρμες ε, σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση και τη συναλλαγή ε, μεταξύ α, των, ε, των διαφόρων παραγόντων, οπότε θα πρέπει εδώ να υπάρχει μια ισορροπημένη αντιμετώπιση αυτών των δύο διαφορετικών διαστάσεων. και μία σειρά από κεντρικούς αντισυμβαλόμενους της Ευρώπης, ε, ειδικότερα οι μεγαλύτεροι, εδώ και ένα χρόνο έχουν ξεκινήσει ακριβώς την προετοιμασία τους ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν ε, και περισσότερα επιχειρησιακά κομμάτια και νομίζω πως ε, σε βάθος χρόνου θα είμαστε σε θέση να έχουμε την κατάλληλη υποδομή η οποία θα μας επιτρέπει να παρέχουμε αυτές τις ε, υπηρεσίες αποτελεσματικά για την ευρωπαϊκή αγορά. Αλλά βέβαια όλα αυτά θα χρειαστούν λίγο παραπάνω χρόνο. Συνοψίζοντας λοιπόν, έτσι όπως έχουν τα πράγματα και έχοντας σε και τις αντιδράσεις απέναντι σε αυτή την πρόταση της ε, ΕΣΜΑ, ε, θεωρώ πως έχουμε επιτύχει με την Επιτροπή ένα καλό επίπεδο ισορροπίας και νομίζω πως θα είμαστε σε θέση αυτό το χρόνο να κάνουμε και τις απαραίτητες διορθώσεις. Ευχαριστούμε. Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Κομπάρη και από το Ρινιού, θέλω να σας υπενθυμίσω σε όλους ότι πρέπει να προσπαθούμε να τηρύνουμε το χρόνο μας, γιατί είναι πολύ δύσκολο να συντονίσω, όπως καταλαβαίνετε, τη συνεδρίαση εξ αποστάσεως, οπότε είναι δύσκολο για μένα να σας υπενθυμίζω πότε έχουν ολοκληρωθεί τα τρία λεπτά, γιατί τότε σας κόβω το λόγο. Οπότε σας παρακαλώ φροντίστε εσείς. Λοιπόν, κύριε Κομπάρικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Καλώς ήρθατε. Η Επιτροπή σας θα πρέπει να φροντίσει ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι από τρίτε χώρες θα τηρούν τις προδιαγραφές, κυρίως όσον αφορά την κατηγορία 2 κεντρικών ε, αντισυμβαλόμενων. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό, μπορείτε να μας πείτε ε, περισσότερο, τι εμπειρία έχετε εσείς που την αναφέρατε εσείς στη ρύθμιση για την σύνταξη του μνημονίου κατανόησης, για παράδειγμα. Και μια ακόμα ερώτηση. Θέλω την άποψή σας για το πώς θα αντιμετωπίσετε δυσκολίες σε συνεργασία με τρίτες χώρες. Για παράδειγμα, πώς θα αντιμετωπίσετε μια κατάσταση όταν μια αρχή τρίτης χώρας είναι απρόθυμη να προσφέρει πληροφορίες πώς θα μπορέσει να κάνει σωστά την αξιολόγησή της η Εποπτική Επιτροπή για τους κεντρικούς αυτούς αντισυμβαλόμενους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απάντηση. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να τηρήσω τα τρία λεπτά. Ναι. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και απαιτούσε μεγαλύτερη απάντηση. Λοιπόν, τώρα, ας πούμε ότι είμαστε υπό το και έχουμε αυτά που αναφέρονται στο ΕΜΙΡ που απαιτεί από τους κεντρικούς συμβαλόμενους να δίνουν κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες, να συμμορφώνονται στους κανόνες μας και να, δέχονται τα, να συμμορφώνονται με τα μέτρα τα οποία εμείς επιβάλλουμε. Αυτό υπάρχει. Τώρα, μια οντότητα η οποία βρίσκεται σε τρίτη χώρα, βρίσκεται σε μια άλλη νομική δικαιοδοσία και πρέπει κανείς να μπορεί να πάει, να έχει πρόσβαση στην ενημέρωση, στις πληροφορίες και σίγουρα χρειάζονται κάποιες διατάξεις από αυτού. Οι διαδικασίες τώρα βάσει των οποίων μπορείτε να συλλέξετε πληροφορίες και αυτές είναι ένα θέμα γιατί υπάρχουν πολλά διαφορετικά ε, ξένα νομικά συστήματα όπως είναι διαφορετικό και εκείνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν πώς συλλέγονται τα δεδομένα φάση των ε, τοπικών διαδικασιών. Ό,τι προβλέπει η διαδικασία της τρίτης χώρας. Εδώ έχουμε να κάνουμε πολλά διαφορετικά νομικά συστήματα. Υπάρχει δηλαδή καταρχήν το τοπικό σύστημα που ρυθμίζει τα περισσότερα και υπάρχει βέβαια και το ΕΜΙΡ. Στην πράξη τώρα τι κάνεις. Ε, προσπαθούμε να συζητήσουμε με τον τοπικό ρυθμιστή για να συζητήσουμε τη συγκεκριμένη περίπτωση, να πούμε τι μας ενδιαφέρει. Αν πρόκειται για θέμα συμμόρφωσης, είναι πολύ σημαντικό να έχεις και απόρριτες πληροφορίες από τον εθνικό ρυθμιστή. Ή και αυτό έχω κάνει εγώ στην προσωπική μου εμπειρία για την εποπτεία επιχειρήσεων. Προσπαθούμε από κοινού να συνεργαστούμε. Είναι πολύ σημαντικό η συλλογή των πληροφοριών να γίνεται με τους σωστούς κανόνες. Για τελείως είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις χρησιμοποιήσει κανείς αν προχωρήσει σε προσφυγή. αν οι δραστηριότητες του κεντρικού αντισυμβαλόμενου από τρίτη χώρα που δρά στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικές, ε, τότε φυσικά και πρέπει να υπάρχει ο σωστός έλεγχος, αλλά χρειάζονται πληροφορίες για να μπορέσει η εποπτική αρχή να προχωρήσει στην εποπτεία και να επιβάλλει συμμόρφωση. Να επιβληθούν κυρώσεις, ό,τι άλλο χρειάζεται, που προβλέπεται στο ΕΜΙΡ. Έμεινα στα τρία λεπτά που μου ζητήσατε. Άμα θέλετε περισσότερα, ευχαρίστω. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ. Ξέρω, μερικέ φορέ είναι δύσκολο να απαντήσει κανεί σε τρία λεπτά. Γιατί οι ερωτήσει είναι πολύ ενδιαφέρουσε και απαιτούν περισσότερο χρόνο, αλλά έχουμε περιορισμένο χρόνο. Τι να κάνουμε. Στο τέλο, στα συμπεράσματα θα μπορούσατε να προσθέσετε κάτι αν θέλετε. Ο Αντώνιο Ρινάλντι τώρα, ID. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε την άλλη. Αξιότιμη κυρία Νικολέτα Τζούστο, χαίρομαι που καλύπτεται το υψηλό προφίλ ε, που απαιτείται σε αυτό το ανώτατο όργανο εποπτείας στην Ιταλία με μεγάλη διεθνή εμπειρία και στην ΕΣΜΑ. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Δεδομένου ότι στο παρελθόν η δράση της ΕΣΜΑ ε, στο εσωτερικό της για συντονισμό υπήρξε μικρή ελαφριά light. Τώρα η Επιτροπή Εποπτείας τι θα κάνει όσον αφορά τη CCP που θα μπορούσαν να πληρούν όλες τις ε, προϋποθέσεις ε, για να αντισταθούν σε συντονισμούς από εθνικούς οργανισμούς στο πλαίσιο της διασφάλισης των συστημικών κινδύνων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Πολύ ενδιαφέρουσα. Πράγματι το ΕΜΙΡ είναι ένας κανονισμός σχετικά νεαρός. Πριν από το ΕΜΙΡ δεν είχαμε τίποτα για τους CCP στην Ευρώπη. Όπως είπα στην εισαγωγή μου, έχω προεδρεύσει την ε, Επιτροπή της ΕΣΜΑ Έχω εμπλακεί στον καθορισμό των μέτρων υλοποίηση για το ΕΜΙΡ 1, αλλά έχω συμμετάσχει και στο συντονισμό των εποπτικών πρακτικών. Η CCP είναι πολύ και διαφορετική σε μέγεθος, σε πολυπλοκότητα δραστηριοτήτων, επίπεδο ε, διεθνούς δραστηριότητας, εξυπηρετούν ε, διάφορους τύπους πλατφορμών και έτσι είναι πολλοί και διαφορετικοί και χρειάζονται πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις. Αλλά η CCP είναι αλληλένδετη, οπότε ο κίνδυνος ε, του να δημιουργηθούν προβλήματα χωρίς να είναι απαραίτητα λάθος των CCP λόγω, ακόμα και αν ε, έχουν μικρό μέγεθος μπορούν να δημιουργήσουν λόγω του ότι είναι αλληλένδετοι προβλήματα. Έτσι λοιπόν υπάρχει ανάγκη να υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας για να διασφαλιστεί το σύστημα, να προστατευτεί από συστημικούς κινδύνους. Εμείς ε, ξεκινήσαμε ήδη ε, αξιολογήσεις μεταξύ ομοτήμων, stress test και τώρα η ΕΣΜΑ έχει φτάσει στο τρίτο επίπεδο stress test, το EMIR 2, επισημοποιεί αυτή τη στιγμή, θεσπίζει στο κανονιστικό πλαίσιο διάφορα βήματα τα οποία διασφαλίζουν το συντονισμό. Πρώτα απ' όλα διάφορες ε, δράσεις ε, ε, αφορούν την οργάνωση του CCP, οργάνωση εντός της οποία απαιτείται μια γνωμοδότηση του οργάνων συντονισμού και αυτό ενισχύει το ρόλο του συντονισμού, το συντονιστικό ρόλο, χωρίς να αρνούμαστε ότι Σε τελική ανάλυση η τελική ευθύνη είναι της ρυθμιστικής αρχής ε, της ε, οικίας χώρας. Θα υπάρχουν ωστόσο ισχυρά μηνύματα από την Επιτροπή η μπορεί να ζητήσει και από το ΕΣΜΑ να εκδώσει γνωμοδοτήσεις, συστάσεις, βήματα τα οποία θα απαιτήσουν κάποια επίσημη δράση ουσιαστικά από, τον, ε, από τη ρυθμιστική αρχή της οικίας χώρας. Η σχέση, οι σχέση αυτές ε, με τα όργανα, τα κολέγια τα οποία επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών για πολύ συγκεκριμένα CCP, ε, με συμμετοχή όλων των αρχών που ελέγχουν αυτό το CCP και με τη συμμετοχή της ΕΣΜΑ, αυτό ο ρόλος θα παίξει ε, σημαντικό ρόλο, θα αποτέλεσε ένα επιπλέον εργαλείο που θα βελτιώσει το ρόλο τη ΕΣΜΑ στο συντονισμό και θα ενισχύσει το συντονισμό αυτό. Θα ήθελα επίση να πω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε σε καμία περίπτωση ότι το EMIR 2.2 με την Εποπτική Επιτροπή CCP λειτουργεί στο πλαίσιο του κανονισμού ΕΣΜΑ που έχει αναθεωρηθεί κάποια δικαιώματα του ΕΣΜΑ που παλιότερα δεν ήταν σαφή. Όταν ξεκίνησε, για παράδειγμα, διάφορε ε, αρμόδιες αρχές απαγόρευαν σε προσωπικό του ΕΣΜΑ ή της Επιτροπής του ΕΣΜΑ να μπουν, να τεθούν σε επαφή, να αποκτήσουν επαφή με CCP για να λάβουν πληροφορίες για stress test, για ε, αξιολόγηση μεταξύ ομοτήμων. Όλα αυτά έχουν αλλάξει τώρα, έχουν διευθετηθεί γιατί τώρα υπάρχει συγκεκριμένοι κανόνες για την ε, συνεργασία μεταξύ ομοτήμων η επαλήθευση, το, το πάνελ επαλήθευσης και ο ρόλος του πάντα ήταν αμφισβητήσιμο. Τώρα θεσπίζεται στις αρμοδιότητες ε, της Εποπτική Επιτροπής του CCP. Αυτό που έχουμε τώρα πιστεύω αποτελεί μια καλή ισορροπία μεταξύ της ανάγκη του να αφήσουμε ε, την οικία αρχή να διατηρεί την κύρια εποπτεία του CCP, CCP και διασφαλίζοντας ένα καλό επίπεδο συνεργασίας και εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα Σβέν Κιγκόλτ από τους Πρασίνους. Yeah, good morning. Thank you. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. λόγω του τεχνικού χαρακτήρα των κεντρικών των και του σχετικού κανονισμού και λαμβάνοντας υπόψη ε, και τη σύνεση που θα πρέπει να επιδεικνύεται σε ό,τι αφορά την επιβολή των κατάλληλων προϋποθέσεων στον τραπεζικό τομέα, σε επίπεδο ESRB και συστημικών τραπεζών και ούτω καθεξής. Πώς α, θεωρείτε πως θα πρέπει να διασφαλιστεί ε, το ότι ακριβώς η, η κανονιστική ρύθμιση για τους ε, κεντρικούς αντισημανόμελους δεν θα περάσει μέσα από αυτό το κάψουλ, δηλαδή αυτήν ουσιαστικά την παγίδευση σε ό,τι αφορά το, το νομοθετικό πλαίσιο για την ανάληψη δράση από την δική σα πλευρά. Έχουμε δει δηλαδή κάτι ανάλογο που είχε γίνει ε, σε επίπεδο EBA, οπότε σας ερωτώ ποια είναι τα μέτρα που θέλετε να αναλάβετε έτσι ώστε να υπάρχει κατάλληλη αποστασιοποίηση από την δική σας πλευρά από τον κλάδο τον οποίο καλείτε ακριβώς να ελέγχετε και τον οποίο καλείστε να, να έχετε την εποπτεία του. Ευχαριστώ, λέει ο ε, ομιλήτρια. Ε, είναι μια πολύ εύστοχη ερώτηση αυτή και δύσκολη να απαντηθεί. Πράγματι έχουμε λοιπόν ε, κάποιους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους οι οποίοι πραγματικά είναι πολύ σημαντικοί στις ε, αγορές μας ε, και οι οποίοι εκτελούν πολύ σημαντικές λειτουργίες. Άρα θα πρέπει να επιτύχουμε την αποφυγή αυτού του regulatory capture, αυτής της παγίδευσης, ας το πούμε έτσι, στο κανονιστικό πλαίσιο. Αλλά νομίζω πως η Εποπτική Επιτροπή για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους θα παίξει εδώ σημαντικό ρόλο γιατί πλέον έχει, όπως αναφέραμε ήδη, ε, την αρμοδιότητα να εξετάσει τις αποφάσεις που θα λαμβάνει η αρμόδια ρυθμιστική αρχή. Με αυτόν τον τρόπο, νομίζω, πως ε, θα έχει την δυνατότητα να κρατάει αυτές τις αποφάσεις ε, και να εξετάζει ακριβώς ε, τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζει εδώ τα πράγματα η Εθνική Καονιστική Αρχή. Δηλαδή θεωρώ πως αν υπάρχει κίνδυνος του regulatory capture, αυτός αφορά περισσότερο στις εθνικές ε, ρυθμιστικές αρχές. Δηλαδή αυτή η Εποπτική Επιτροπή για τους ιατρικούς Συμβαλλόμενους είναι ε, διαφοροποιημένη και από την ίδια την ΕΣΜΑ και το Διοικητικό Συμβούλιο. Δηλαδή πραγματικά πρόκειται εδώ για έναν ε, ξεχωριστό φορέα Έχουμε δηλαδή έναν δικό μα πρόεδρο και έχουμε δύο ανεξάρτητα μέλη και ακριβώς ο στόχος είναι εδώ η ανεξαρτησία. Με στόχο τον έλεγχο και την κατάλληλη αξιολόγηση αλλά και την... να δίνονται και κατάλληλε προειδοποιήσει σε σχέση με τι αποφάσει που λαμβάνονται. Και βέβαια οποιασδήποτε αποφάσεις λαμβάνει αυτή η Αποπτική Επιτροπή για τους ιατρικούς αντισυμβαλόμενους θα πρέπει να λαμβάνει την έγκριση από ε, την ηγεσία της ΕΣΜΑ. Θα δημόσαστε ότι η σχετική πρόφαση δεν είχε γίνει δεκτή ε, από το συνομοθέτηση ό,τι αφορά την ΕΣΜΑ, οπότε νομίζω πως τώρα υπάρχει χαμηλότερος κίνδυνος για αυτό το regulatory capture. Πέραν αυτού υπάρχει μια σειρά από κανόνες ως προς το πώς θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε εναντί του κλάδου σε ό,τι αφορά το ζήτημα του σύγκρουσης συμφερόντων, των σχετικών δηλώσεων που θα πρέπει να υπογράψω και εγώ από τη δική μου ε, πλευρά προσωπικά εάν πράγματι διοριστώ. Hello? Okay. I'm sorry. Ευχαριστούμε. Συγγνώμη, δυσκολεύτηκα να συνδεθώ. Γι' αυτό καθυστέρησα. Τώρα συνεχίζουμε και περνάμε στον κύριο Έπινγκ, ECR. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε. Οι επικρίσεις για την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλόμενων ακούγεται ως να πρόκειται για κάτι εντελώς ε, κενό και που έχει τις επιπτώσεις ε, το αυτό το θέμα και στην αρχή κινητών αξιών και αγορών. Εσείς τι μπορείτε να κάνετε για να το αντιμετωπίσετε αυτό. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Όντω έγιναν πολλές συζητήσεις. Αλλά εγώ δεν θα έλεγα ότι δεν υπάρχει εποπτεία. Πρώτα απ' όλα υπάρχει αυτή η Επιτροπή η οποία αποτελείται από ανεξάρτητα μέλη επίσης. Θα δούμε πώς θα οργανώσουμε τη δουλειά μας με το υπόλοιπο προσωπικό. Πάντως, η δουλειά που θα να φέρουμε σε πέρας θα είναι τεράστια, γιατί τελικά δεν θα πρόκειται μόνο για γενικού περιεχομένου συζητήσεις όσον αφορά την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλόμενων, θα έχει να κάνει και με εκθέσεις προς τα ευρωπαϊκά όργανα, με αποφάσεις για την ε, κύρωση ή όχι και υπάρχουν πολλές δυσκολίες εκεί. Γιατί πρέπει να είμαστε σε θέση να έχουμε πρώτα ε, μία συμβουλή από συμβουλευτικά όργανα ε, προς την Επιτροπή αυτή την εποπτική και μετά να προχωρήσουμε. Ο συνάδελφός σας που πρώτος πήρε το λόγο σήμερα το πρωί τόνισε ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχα συστήματα. Οι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι οι οποίοι θα ταξινομηθούν σε κάποια κατηγορία θα πρέπει να δούμε αν θα έχουν κάποια εξαίρεση ή όχι από συμμόρφωση, ανάλογα βέβαια με την ομοθεσία ΕΜΙΡ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχετε πληροφορίες για τις επιδόσεις, να αναλύσετε αυτές τις επιδόσεις για να μπορέσετε να κρίνετε κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση ή όχι. Μπορεί να χρειάζονται επιπλέον πληροφορίες, άρα αιτήματα να σταλούν στους κεντρικούς θετσιβαλόμενους κλπ. κλπ. Δεν θα έλεγα λοιπόν ότι δεν θα υπάρχει τίποτα. Διαπραγματεύσεις επίσης με τις αρχές των τρίτων χωρών εφόσον χρειάζεται. Κάποιοι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι από τρίτες χώρες που δρούν υπό το καθεστώς εξαίρεσης, παρέκκλησης, υπό τον ΕΜΙΡ 1, για αυτούς που κοινοποιούν περιμένοντας ε, την αντιστοιχία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάτι που παραμένει αναγκαίο. Πάρα πολλές ε, εκτιμήσεις πρέπει να κάνουμε αντιστοιχίας. Υπάρχει το Brexit, ε, υπάρχει το ότι μπορεί να είναι ε, πολύ μεγάλος ο κεντρικός αντισυμβαλόμενος. Υπάρχουν ένα σωρό κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι που δρούν σε τοπικές αγορές υπό το καθεστώς που λέμε και που περιμένουν ακόμα την ισοδυναμία. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ζητάει κανένας άλλος το λόγο από ό,τι βλέπω. Οπότε κυρία Τζούστο, αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δύο λεπτά που έχετε ακόμα στη διάθεσή σας για τα συμπεράσματά σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι η συζήτησή μας και οι ερωτήσεις που μου κάνατε με τις απαντήσεις μου επιτρέπουν να καταλάβετε λίγο πολύ ποιες θα είναι οι προτεραιότητες της Εποπτικής Επιτροπής Κεντρικών Αδεσυμβαλωμένων και ποιος θα είναι ο σημαντικός ρόλος της. Ε, φυσικά αν υπάρχουν επικρίσεις θα δούμε όταν ξεκινήσουμε τις εργασίες μας εφόσον συμμετέχω κι εγώ και εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει η Υποπτική αυτή Επιτροπή όταν θα έχει προχωρήσει θα αρχίσει να ασχολείται με θέματα όπως είναι το Brexit. Αλλά υπάρχουν και πολύ περισσότερα θέματα, υπάρχουν πολλές τρίτες χώρες από τις οποίες έχουμε κεντρικούς τατσιβαλόμενους και πρέπει να τις λάβουμε υπόψη. Είναι τεράστιο το έργο που πρέπει να τελεστεί στην Ευρώπη για να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε ε, σωστή εποπτεία και συγκρίσιμη με τα όσα κάνουμε για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους στην Ευρώπη, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Είναι ένα τεράστιο έργο σε διεθνές επίπεδο. Παίζουν τεράστιο ρόλο οι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι στα παράγωγα, μεταξύ άλλων τα όσα λέει το G20 επίσης, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες πολύ σημαντικοί για τα μετοχικά κεφάλαια, για την για το κανονιστικό πλαίσιο όλων αυτών. Και εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε όλα να προχωρήσουν ομαλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάλι κυρία Τζούστο και όλα τα μέλη για τις ερωτήσεις. Ας κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα δύο λεπτών για να δώσουμε το χρόνο στην επόμενα υποψήφιο να συνδεθεί. Και εγώ εδώ θα εγκαταλείψω την Προεδρία της Ακρόασης και θα τη δώσω στον κύριο Έπινγκ, τον Αντιπρόεδρο, τον οποίο ευχαριστώ για τη διαθεσιμότητα που έδειξε. Ευχαριστώ πολύ. morning, Miss Vent. We... Καλημέρα κυρία Βέντ, μπορείτε να πατήσετε το speak για να δοκιμάσουμε τη σύνθεσή σας. Good morning. Καλημέρα. Με ακούτε, σας ακούμε και σας βλέπουμε. Ευχαριστώ. Well, colleagues, let's uh, resume the, the... συνεχίσουμε την συνεδρίαση και καλωσορίζω την κυρία Φρούκελιν Βέντ. Ελπίζω να μας βλέπει. Να ζητήσω πρώτα απ' όλα συγγνώμη για το χρόνο. Διότι έχει συνδεθεί από την Washington, όπου αυτή τη στιγμή είναι 4 και 20 το πρωί, τη νύχτα. Οπότε ας είμαστε επίοικείς μαζί της και να μην την πιέσουμε πολύ. Γιατί είναι λίγο νωρί για αυτή. Είναι, είναι υποψήφια για μία από τι δύο θέσει των αναξαρτητών μελών τη Νέα Εποπτική Επιτροπή ε, για κεντρικού αντισυμβολωμένου. Η ΕΣΜΑ ειδοποίησε το στις 27 Αυγούστου το Κοινοβούλιο για την απόφαση επιλογής της κυρίας Βουέντα από έναν κατάλογο τελικών υποψηφίων για ανεξάρτητο μέλος του της Εποπτικής Επιτροπής μετά από τη δημοσίευση των κενών θέσεων το 2019 και μετά από μια επιλογή ανοιχτή. Ξέρετε πώς οργανώνεται απόψη χρόνων αγορητών η συνάντηση. Πέντε λεπτά η εισαγωγή της κυρίας Βέντ, ερωτήσεις μετά και απαντήσεις για τέσσερα λεπτά κάθε φορά, ένα λεπτό για την ερώτηση, τρία για την απάντηση. Κάθε πολιτική ομάδα έχει μία χρονοθυρίδα. Εάν το επιτρέψει ο χρόνος θα δώσουμε και άλλες χρονοθυρίδες βάσει διαδικασίας Catch the Eye, λαμβάνοντας υπόψη το βάρος της κάθε πολιτικής ομάδας. Στο τέλος θα καλέσω την κυρία Βέντ να κάνει μία τελική ε, παρουσίαση δύο λεπτών. Το πολύ. Ας δώσουμε το λόγο τώρα στην κυρία Γουέντ για πέντε λεπτά για να μας κάνει μια εισαγωγή. Καλημέρα από την Washington DC. Πράγματι είναι τέσσερις και είναι λίγο σκοτεινά εδώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους σας που μου δίνετε την ευκαιρία να σας μιλήσω και να σας κάνω αυτή την παρουσίαση. Είναι τιμή που μιλώ σε εσάς τους αιρετούς εκπροσώπους ε, των Ευρωπαίων λαών ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αντιλαμβάνομαι πόσο δημόσιο ρόλο και σημαντικό έχει η Εποπτική Επιτροπή ε, σε θέματα εποπτείας. Όλη η οικονομική σταθερότητα, η προστασία των πολιτών, ε, των επενδυτών και η ενίσχυση των κεφαλαγορών εξαρτώνται από αυτήν. Και εσείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχετε λάβει πολύ σαφή ε, ε, και μεγάλες αποφάσεις με το ΕΜΕΡ 22 που ενισχύει την εποπτεία και την βελτιώνει και χαίρομαι που βρίσκομαι στο δικό σα τελικό κατάλογο υποψηφίων και φιλοδοξώ να εργαστώ με μεγάλο πάθος αυτή την Εποπτική Επιτροπή αν με εξουσιοδοτήσετε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τον ε, τελευταίο κανονισμό για τον οποίο ε, υπήρξε μια συμφωνία ε, πριν το καλοκαίρι για το COVID και ήταν μεγάλο επίτευγμα. Όλη μου η σταδιοδρομία αφιερώθηκε στην ενίσχυση των κεφαλαίων και των σχετικών δομών. Εγώ ξεκίνησα στο Γιονέξτο, οπότε γνωρίζω τον ιδιωτικό τομέα. Μετά πέρασε στην Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα όπου επόπτευα CCP και την τελευταία δεκαετία ηγούμε ε, πολυπολιτισμικών ομάδων στην αξιολόγηση CCP σε ολόκληρο τον κόσμο. Φιλοδοξώ λοιπόν να, φέρω, να συνεισφέρω με αυτές τις τεχνικές γνώσεις και αυτές τις διπλωματικές εμπειρίες, την πολιτική ευαισθησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το καλό των Ευρωπαίων πολιτών. Από αυτή την άποψη έχω τρεις φιλοδοξίες. Η πρώτη μου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας ε, ε, μεταξύ ΕΣΜΑ και εσάς, μεταξύ της Εποπτικής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων ευρωπαϊκών οργάνων. Μια Εποπτική Επιτροπή πιστεύω θα μπορέσει να είναι επιτυχής στο ρόλο της μόνο αν καταλάβει τον ρόλο της μες στο ευρύτερο οικοσύστημα και πράγματι η Επιτροπή για να είναι ανεξάρτητος επόπτης πρέπει να καταλάβει ότι ανεξάρτητος δεν σημαίνει απομονωμένος Και γι' αυτό η πρώτη μου φιλοδοξία είναι να έρθω σε επαφή με εσά, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να συζητήσω μαζί σας για να καταλάβω τι είναι σημαντικό για εσάς, Τι σας ανησυχεί, τι φοβάστε όσον αφορά τους CCP, αλλά και τα σχετικά ζητήματα όπως η, η φόρο ε, οικονομία. Η δεύτερη μου φιλοδοξία είναι να χτίσω γέφυρες μεταξύ των εποπτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με γνώμονα ένα σημαντικό στόχο που έχουμε αποφασίσει να προωθήσουμε την εποπτική σύγκληση. Ξέρω από πρώτο χέρι ότι δεν είναι πάντα εύκολο, χρειάζεται χρόνο. Όταν εργαζόμουν στην Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα ως επόπτης, Ε, συζήτησα μνημονία και με άλλους επόπτες ε, και ε, κλασικά στην αρχή υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης και τα πράγματα δεν είναι εύκολα αλλά με τα χρόνια χτίζεται αυτή η εμπιστοσύνη οικοδομείται μεγαλύτερη εκτίμηση και αρχίζει η εργασία να γίνεται πιο αποτελεσματική μερικές φορές αυτές οι εποπτικές αρχές αποτελούνται από πολλές διαφορετικές αρχές μπορεί να είναι και έτσι λοιπόν η δεύτερη μου φιλοδοξία για την ε, Εποπτική Επιτροπή CCP είναι να το καταλάβουμε και αυτό. Και η τελευταία μου φιλοδοξία και όχι λιγότερο σημαντική είναι η προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πιθανές ε, ζημίες λόγω CCP τρίτων χωρών. Και όλοι ξέρουμε ότι με τον Brexit κάποια ε, από τα μεγαλύτερα CCP θα βρεθούν τώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό και το EMIR 2.2 μας δίνει πολλά εργαλεία για την ε, αξιολόγηση, αποτίμηση των CCP, για τον εντοπισμό των κινδύνων και τον μετριασμό τους. Κατά την άποψή μου αυτό θα γίνει αφενός με το να είμαστε αξιόπιστοι αντισυμβαλόμενοι ε, ομόλογοι των CCP τρίτων χωρών, ούτω ώστε να έχουμε τη συνεργασία που είναι αναγκαία και την εμπιστοσύνη που είναι αναγκαία, αλλά επιπλέον ε, αυτή τη σχέση θα δείξουμε ότι ε, θα είμαστε σκληροί εκεί όπου απαιτείται, χωρίς να διατρέχουμε κίνδυνο για τις δικές μας τράπεζες, για, για τα δικά μας συστήματα. Αυτός ο συνδυασμός διπλωματίας με σκληρότητα είναι κάτι που έχω χρησιμοποιήσει επιτυχώς ε, για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όταν αξιολογούσα, αλληλεπιδρούσα και διαπραγματευόμουν με αρχές από ολόκληρο τον κόσμο. Θα ήθελα λοιπόν ε, να συνεισφέρω έτσι στην Εποπτική Επιτροπή CCP της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ ολοκληρώνεται η εισαγωγή μου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και προς το κόνο έχουμε μια καλή ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Βέντε που συνέστε μαζί μας από τη Ουάσιγκτον. Περνάμε τώρα στις ε, ερωτήσεις και απαντήσεις. Καταρχήν η κυρία Ντανούτα Χούμπνερ εκ μέρου του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σας ε, κυρία Βέντε και χαίρομαι που σας ξαναβλέπω εδώ. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα το οποίο είναι το εξής. Ε, ποια θεωρείτε πως είναι η υποδομή εξοπλισμός που έχουν οι αρμόδιοι για την εποπτεία σε ό,τι αφορά τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους. Είναι δηλαδή σε θέση με αυτόν τον εξοπλισμό να παρακολουθούν και να αξιολογούν ε, τους κινδύνους, τους χρηματοπιστωτικούς και της ε, ε, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Επίσης εδώ να αναφέρω ότι τον, ε, τον Ιούνιο το Συμβούλιο του Συστημικού Ρίσκου, κινδύνου δηλαδή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξέδωσε κάποιες ε, συστάσεις σε ό,τι αφορά τα αντιρρήματα, τις ρόλους και το, ε, ε, τα cliff edge, τις επιπτώσεις cliff edge effects, δηλαδή σε ό,τι αφορά το, τα, τις ανάγκες μελλοντικής ρευστότητας, το stress testing και ό,τι καθεξής. Και υπάρχουν βέβαια και τα διεθνή πρότυπα για την μείωση της κλικότητας και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, ε, θεωρείτε πως υπάρχει αυτή η ετοιμότητα από την πλευρά των αρμόδιων για το κανονιστικό πλαίσιο και των εποπτών ε, των κεντρικών αντισυμβαλόμενων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Βέντε, έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χούμπνερ για το ερώτημά σας για τη δυνατότητα που μου δίνετε να αναφερθώ λίγο περισσότερο στις αρμοδιότητες που θα έχουν πλέον οι, ε, οι επόπτες ε, του, για τους κεντρικούς υπό τον κανονισμό ΕΜΕΡ. Το ΕΜΕΡ δηλαδή, εφαρμόζει ένα είδος αναλογική ε, προσέγγισης σε ό,τι αφορά του σχετικού αντισυμβαλόμενους σε τρίτων χωρών. Δηλαδή κάνει μια διάκριση ανάμεσα σε ένα και δύο. Οπότε να απαντήσω ε, σε δύο σκέλη στο ερώτημά σα. Ε, δηλαδή, καταρχήν σε ό,τι αφορά του κεντρικού αντισυμβαλόμενου εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά σε ό,τι αφορά του κεντρικού αντισυμβαλόμενου εντό τη Ένωση. Άρα, λοιπόν, σε ό,τι αφορά εκείνου τρίτων χωρών, έχουμε αυτή την διαφοροποίηση ανάμεσα σε ένα α, και δύο. Δηλαδή, εκείνου που είναι περισσότερο σημαντικοί και λιγότερο σημαντικοί από συστημική πλευρά. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή του οι επόπτε των κεντρικών αντισυμβαλόμενων. Εάν είμαι δηλαδή αξιολογητή από πλευρά ΑΕΜΕΦ και ε, εξετάζω αυτά τα εργαλεία, ναι, θα συμπεράνω ότι πραγματικά είναι επαρκή, ειδικότερα σε ό,τι αφορά του CCP τη ε, πρώτη κατηγορία. Δηλαδή γίνεται χρηματική αξιολόγηση, γίνεται ε, ε, συνομιλία με αυτούς τους ε, CCP. Μπορεί να υπάρξει και μόνο κατανόηση MOU e προκειμένου ακριβώς να αναγνωριστούν κίνδυνοι και ανάπτυξη των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον, την δεύτερη κατηγορία, των, αυτών των των χωρών, ε, εκείνων δηλαδή που είναι συστηματικά πιο σημαντικοί, έχουμε ένα ολόκληρο εύρο εργαλείων. Ε, υπάρχουν δηλαδή ακόμα και επιτόπιε επιθεωρήσει οι οποίε ε, προβλέπονται με τη δυνατότητα επιβολής προστήμων και ούτω καθεξή. Μετά σε ό,τι αφορά μια τρίτη αν θέλετε κατηγορία τη συμβαλόμενη, δηλαδή εκείνος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ βέβαια προφανώ οι Εθνικέ μυθιστικέ αρχέ είναι οι αρμόδιε, αλλά από εκεί και μετά έχουμε και εμεί τα κατάλληλα εργαλεία στη διάθεσή μας. Τώρα, το ερώτημα σας ήταν κατά πόσο ε, θεωρώ ότι αυτά τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι επόπτες των κεντρικών αντισυμβαλόμενων, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά φαινόμενα προκυκλικότητας και ούτω καθεξής. Ναι, εγώ θεωρώ πως αυτά τα εργαλεία επαρκούν. Παρ' όλα αυτά να πω ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται αυτά τα εργαλεία με τρόπο ο οποίος να απηχεί ε, το βαθμό κατανόησης ακριβώς των κινδύνων, δηλαδή να είναι προσαρμοσμένη η εφαρμογή αυτών των εργαλείων στο είδος των κινδύνων. Δηλαδή σε ό,τι αφορά αυτό το ε, ε, ε για παράδειγμα, ε, η κρίση με το COVID κατέδειξε ότι Ε, είδαμε ότι εδώ λοιπόν ε, μπορεί να υπάρξει ε, επιβάνηση σε ό,τι αφορά την, το, το stress. Οπότε σε επίπεδο εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλόμενων εγώ από τη δική μου πλευρά θα ταχθώ υπέρ της βελτίωσης του τρόπου με τον οποίο αντιδρούν σε τέτοιου είδους εκκρίσεις οι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι. Δηλαδή από τη μία πλευρά αξιολόγηση των κινδύνων, αλλά από την άλλη πλευρά ο ρόλος των ε, οι οποίοι αντιμετωπίζουν και αυτά τα ζητήματα ρευστότητα. Επίσης, θεωρώ πώ υπάρχει πλέον βάση ε, για να εξετάζουμε όχι μόνο τους συλλητικούς αντισυμβαλλόμενους αλλά και τους συμμετέχοντες στην αγορά, τους ε, παίκτες δηλαδή στην αγορά σε ό,τι αφορά το πλαίσιο ρευστότητα. Ε, δηλαδή θα πρέπει να εξετάζονται χωρίς όμως να περιλαμβάνονται στο εύρος αρμοδιοπτήτων εποπτείας από την πλευρά των, των κεντρικών αντισυμβαλλόμενων Ευχαριστούμε. Περνάει και ο χρόνος. Να τηρείτε το χρόνο σας, υπενθυμίζω, λέει ο Πρόεδρος. Δεύτερος ομιλητής, η κυρία Εύελιν Ρέγνερ, Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ. Καλή μέρα, βέβαια πολύ πρωινή καλημέρα. Εγώ θέλω να ρωτήσω για την επίφαση της πράσινης διάστασης. Είναι πολύ σημαντικό να μην μπερδευόμαστε όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Κατά τη γνώμη σας, λοιπόν, η ποιότητα και το κριτήριο το κατά πόσο είναι πράσινη ή όχι μια επένδυση πώς ε, μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό του greenwashing, της επίφασης δηλαδή ότι κάτι είναι οικολογικό και πράσινο. Ελπίζω ότι θα υπάρξουν πολύ σύντομα οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα πράσινα ομόλογα, οπότε εν ώψη αυτού ε, ρωτάω και θέλω να ξέρω τι πιστεύετε. Απάντηση για τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας αυτή. Πράγματι, Οι πράσινες επενδύσεις είναι ένας πολύ σημαντικός ε, στόχος και για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Νομίζω ότι όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ε, θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα με μεγάλη προτεραιότητα στην πολιτική τους. Το θέμα του greenwashing, της πράσινης επίφασης, όπως είπαμε νωρίτερα, είναι κάτι που δεν έχει να κάνει ακριβώς με το συμψηφισμό και τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους. Είναι όμως ένα σημαντικό ζήτημα και πιστεύω ότι όσον αφορά τον κεντρικό συμψηφισμό θα έπρεπε να τονίζουμε πιο πολύ ε, τα βιώσιμα χρηματοπιστωτικά. Και αναφέρεται και για τους κεντρικούς ενσυμβαλόμενους ότι θα πρέπει να κάνουν δοκιμές αντοχής. Από μια μεριά υπάρχει το λειτουργικό σκέλος που πρέπει να προστατεύεται και από την άλλη μεριά υπάρχουν οι φυσικοί πόροι από τους οποίους έμεσα μπορούν να αποφεληθούν οι επενδυτές. Αλλά πρέπει να δούμε μήπως υπάρχει υπερβολική έκθεση σε κάποιους τομείς που δεν είναι πράσινοι. Πιστεύω ότι η CCP και η ΕΣΜΑ στο δικό του χώρο καθένας μπορούν να συνεισφέρουν υπέρ βιώσιμων χρηματοπιστωτικών υπέρ των Ευρωπαίων επενδυτών και Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε. Renew. Η κυρία Κάρολάιν Νάχτεραλ, η οποία βρίσκεται, θα συνδεθεί εξ Ένα λεπτό ερώτησή σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω κάποιες ερωτήσεις για σας. Στην εισαγωγή σας ήδη αναφερθήκατε στην Συμφωνία για την Ανάκαψη και την Εξυγίανση των CCP. Πολλοί από αυτούς υποστηρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο οι Ευρωπαίοι ε, κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους αντίστοιχους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένης λοιπόν της εμπειρίας που εσείς διαθέτετε και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εσείς πώς ε, βλέπετε αυτόν τον ισχυρισμό και ποιες θα είναι οι κύριες δυσκολίες που θα έχουν να αντιμετωπίσουν την επόμενη δεκαετία οι Ευρωπαίοι ΣΥΣΥΠΙΣ. Και τέλος, αναφερθήκατε στην τρίτη σας φιλοδοξία. Θέλω να ξέρω, ο ρόλος της ε, Εποπτικής Επιτροπής και των Κεντρικών Αντισυμβαλόμενων ποιος θα είναι εν με το Brexit και τι θα γίνει με τους κεντρικούς Αντισυμβαλλόμενους που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πώς θα φροντίσουμε να υπάρχει συνέχεια στην, στις δραστηριότητε τους. Ευχαριστούμε. Απάντηση για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω. Ναι. Ε, να σας ε, καθησυχάσω με το εξή. Όταν πρόκειται για την ανάκαψη και την εξυγίανση, πράγματι έχουν γίνει κάποιες επιλογές στη διαδικασία προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα πολιτικό συμβιβασμό και να καλυφθούν όλες οι πλευρές. Το κείμενο, αυτό για την ανάκαψη και την εξυγίανση, βασίζεται σε διεθνείς προδιαγραφές. Αυτό μας καθισκάζει κάπως όσον αφορά την ισότιμη ε, αντιμετώπιση. Αλλά, όπως λέτε κι εσείς, υπάρχουν κάποιες διαφορές που ίσως καταλήξουν σε διαφορετικές συνθήκες και άνηση κατάσταση. Πάντως, οι διαφορές αυτές πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα διαφορετικά συμφέροντα των CCPs, των συμψηφιζόμενων. Ε, όλα αυτά καταλήγουν σε διαφορόπους και διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ουσιαστικά πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους. Έτσι θα είναι ισχυρό το σύστημα. Από την άλλη μεριά, όπως λένε οι ίδιοι οι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι, χρειάζεται παραπάνω κεφάλαιο ε, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, κάτι το οποίο μπορεί να τους οδηγήσει σε μειονεκτική θέση απέναντι στους αντίστοιχους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τελικό κείμενο δεν ζητάει βέβαια επιπλέον κεφάλαιο, αλλά ζητάει κάποια εγγύηση. Όχι κεφάλαιο έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ. Για μένα λοιπόν είναι μια απόλυτα λογική προσέγγιση για ε, κάποια δικαιοδοσία η οποία βασίζεται σε διεθνείς προδιαγραφές αλλά βέβαια η κάθε δικαιοδοσία καλείται να κάνει κάποιες επιλογές. Πάντως έχουν εναλλακτική για την ανάλυση κινδύνου οι CCPs, από την άλλη μεριά πρέπει να καθισχαστούν ότι δεν υπάρχει άνηση αντιμετώπιση. Αυτά για την πρώτη σας ερώτηση. Η δεύτερη ερώτησή σας ήταν για τις κύριες προκλήσεις, αν σας κατάλαβα καλά, που θα αντιμετωπίσουν οι κεντρικές συμβαλόμενοι συμμορφόμενοι προς τον κανονισμό για την ανάκαμψη και την εξυγένση. Από τη δικιά μου εμπειρία, οι περισσότεροι κεντρική συμβαλόμενοι, αν όχι όλοι, ήδη έχουν ένα σχέδιο ανάκαμψης. Γιατί το ζητά αυτό, το ζητούν οι διεθνείς προδιαγραφές. Ο κανονισμός βέβαια εφαρμόζεται μετά από κάποιους μήνες. Αντιμετωπίζουν το θέμα ε, του να επανεξετάσουν, να δουν τις αδυναμίες, τα ισχυρά σημεία του σχεδίου τους ανάκαμψης προκειμένου να το ευθυγραμμίσουν με τις νέες απαιτήσει. Αυτό μπορεί να είναι μια δυσκολία. Εγώ προσωπικά και έχω διαβάσει τις απαιτήσει και πολύ χάρηκα που βλέπω ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ότι αποτελούν μέρος μιας γενικότερης ομάδας ε, παραγόντων. Γιατί μερικέ φορές οι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι κοιτάνε μόνο το δικό του τον κίνδυνο, τα δικά του τα περιθώρια και δεν συνειδητοποιούν ότι υπάρχει αλληλεσύνδεση με άλλους κεντρικούς αντισυμβαλόμενου και ότι από εκεί κινδυνεύει ε, η, η δουλειά του όλων. Ενώ τώρα νομίζω ότι το καταλαβαίνουν σιγά σιγά. Οπότε το θέμα της ανεξαρτησίας διακόπτει ο πρόεδρος. Πρέπει να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Δίνω λοιπόν το λόγο. Ε, δίνω το λόγο ε, στο, στην πολιτική ομάδα ID, αλλά δεν βλέπω κάποιον ομιλητή ο οποίος ε, έχει καταχωρηθεί. Οπότε περνάμε στους πρασίνους. Σφεν Κίγκος, για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω κύριε Βέντ. Η δική μου ερώτηση είναι αρκετά ευθεία. Ε, ε με τις αρχικές σας δηλώσεις ότι αφιερώσατε τον επαγγελματικό σας σερβίο στην ε, ε, ισχύ αυτών των φορέων, αλλά τώρα ε, στο πλαίσιο μιας εποπτικής αρμοδιότητας θα πρέπει να έχετε περισσότερη απόσταση από εκείνους τους οποίους θα ελέγχετε δημοσίως. Άρα λοιπόν το ερώτημα που για μένα ανακύπτει είναι το εξής. Ε, πώς θέλετε να αποφύγετε το regulatory capture, δηλαδή αυτή την παγίδευση αν θέλετε σε κανονιστικό επίπεδο γιατί μιλάμε για μια σχετικά μικρή κοινότητα αν θέλετε ε, βλέπετε πως ε, ε, οι τράπεζες για παράδειγμα χρηματοπιστωτικοί φορείς είναι πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τέτοιων κανόνων στις δικές τους τράπεζες οπότε Πώ θέλετε να διασφανίσετε ότι δεν θα βιώσουμε κάτι τέτοιο, αυτό το regulatory capture και μέσω αυτών των εποπτικών δραστηριοτήτων για τους κεντρικού αντισυμβαλόμενου από την πλευρά Ευχαριστώ για αυτό το πολύ σημαντικό ερώτημα. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε ότι έχουμε να κάνουμε μια μικρή κοινότητα εντό εισαγωγικών. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι είναι αδύνατο κανεί να κρατήσει τι αποστάσει που χρειάζεται. Όπω γνωρίζετε, αυτή την ε, περίοδο ε, εργάζομαι για το IMF, ε, το Διεθνές Σωματικό Ταμείο, το οποίο έχει ακριβώς πολύ ε, αυστηρούς κανόνες σε σχέση με αυτό το τομείο και γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή το να μπορεί κανείς να χαίρει απόλυτης αμεροληψίας και να μην Ακριβώς ε, ε, λαμβάνει η χώρα αυτό το regulatory capture. Δηλαδή φροντίζω πάντοτε να είμαι ανεξάρτητη και να είμαι σε θέση να αναγνωρίζω κινδύνου, οι οποίοι μπορούν να, να ε, θέσουν αμφίβολο την χρηματική σταθερότητα. Αυτή είναι η δική μου στάση αν θέλετε, αλλά από εκεί και μετά πώς μπορώ να εφαρμόσω κάτι τέτοιο πρακτικά. Ε, με ρωτήσατε. Υπάρχουν μια σειρά από τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να το επιτύχει. Έχω ενημερωθεί σε σχέση με τις πολιτικές της ΕΣΜΑ και το ζήτημα των, των πολιτικών για τη σύγκρουση συμφερόντων και προφανώ είμαι απόλυτα διατεθειμένη να συμμορφωθώ με όλε αυτέ τι προποθέσει, οι οποίε ε, πραγματικά είναι ορθές και ευθυγραμμίζονται πλήρω με την δέουσα συμπεριφορά και τα όσα απαιτούνται. Αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο. Από εκεί και μετά σε ό,τι αφορά ένα, ε, το δυνητικό φαινόμενο των revolving doors, δηλαδή το να αναλαμβάνει κανείς ε, διαφορετικά καθήκοντα ε, στο πλαίσιο ακριβώς του ίδιου κλάδου, με ενδεχομένω σε θέσεις οι οποίες να έχουν αντικρώμενα μεταξύ τους συμφέροντα. Ναι, είναι μια μικρή κοινότητα, αλλά εγώ γνωρίζω πάντοτε σε σχέση με όλες τις θέσεις που αναλαμβάνω ποια είναι τα όρια και ποιες είναι οι υποχρεώσεις και αυτό θα κάνω και στην περίπτωση που διοριστώ εδώ. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά το ε, revolving doors, αυτό το φαινόμενο δηλαδή, ε, το να ε, υπάρχει ο κίνδυνος δηλαδή να χαμηλώσει κανείς αν θέλετε το επίπεδο αυστηρότητας σε ό,τι αφορά τις εποπτήσεις τους δραστηριότητες προκειμένου να λάβει μια άλλη θέση εργασίας σε αυτό το τομέα στο μέλλον είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα επιζήμιο και με βρίσκει απόλυτα αντίθετη. Νομίζω πως ε, το ε, ε, ψήφισμα το οποίο υιοθετήθηκε και νωρίτερα φέτος είναι κάτι που θα πρέπει να επενέσω. Κάτι ακόμα που θα ήθελα να πω είναι ότι κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων σε αυτό το τομέα είναι πολύ σημαντική διαφάνεια. Από ό,τι γνωρίζω η ΕΣΜΑ ακολουθεί μια διαδικασία με βάση την οποία οποιαδήποτε συνάντηση μεταξύ, για παράδειγμα, του Προέδρου αυτής της Εποπτικής Επιτροπής αλλά και φαντάζομαι και ε, μελών ε, της Επιτροπής ε, και άλλων εκπροσώπων των κεντρικών αντισυμβαλόμενων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΣΜΑ και πρόκειται δηλαδή για πολύ σωστές πρακτικές που ταυτόχρονα όμως μας επιτρέπουν να βρισκόμαστε και σε επαφή με, με τον τομέα. Γιατί βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό ως τέτοια υποπτική αρχή να μην ε, δρούμε ε, απομονωμένα από τον ευρύτερο τομέα. Ελπίζω να απάντησα στο ερώτημά σας. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω τώρα το λόγο στο ECR. Δηλαδή, εγώ ο ίδιος παίρνω το λόγο. Το λόγο τώρα στο ECR, δηλαδή στον εαυτό μου και θα ήθελα να απαντήσετε την εξής ερώτηση. Ποιον θα καλέσουν οι, Ευρω... σε περίπτωση κρίση στην Εποπτική Επιτροπή CCP ή τους επόπτες ε, από την Parfait τη Bank de France. Αφού είστε στη Washington, ε, έχει εσείς την επιλογή. Η φιλοδοξία μου είναι ότι αν υπάρχει κρίση με το CCP τον ΗΠΑ θα παίρνουν σε μας. ή τουλάχιστον εμάς. Ε, θα πρέπει να ενημερώνουν και άλλους ε, και άλλες αρχές, αλλά σε κάθε περίπτωση και εμάς. Όπως αναμένουμε θα είναι στις επικατηγορίας 1, τον είπα. Και η φιλοδοξία μου είναι να είμαστε σε τακτική επαφή μαζί τους, ούτω ώστε να καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι συμβαίνει στη ΣΥΠΑ, ότι σε περίπτωση κρίση, ένα από τα πρώτα πράγματα αφού το συζητήσουν εσωτερικά θα είναι να καλέσουν εμά ώστε να μπορούμε να εξελογήσουμε τι ζητήματα υπάρχουν, τι πιθανέ λύσει ε, γίνονται και να λάβουμε μέτρα. Ελπίζω αυτό να απαντά την ερώτησή σα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα κανονικά θα περνούσα στην ΚΟΕ, αλλά η ΚΟΕ δεν βρίσκεται εδώ, δεν έχουμε όνομα στο κατάλογο. Δεν ζήτησε κανείς ε, ε οπότε δίνω το λόγο στην κυρία Βουέντε για δύο λεπτά για να κλείσει την παρουσίασή της. Κλείνοντας ε, αυτό το δύο δεν θα σπαταλήσω πολύ από το χρόνο σας, αλλά ήθελα να σας ευχαριστήσω ξανά που με καλέσατε εδώ για να συμμετάσχω στη συζήτηση αυτή. Ήταν πολύ καλή συζήτηση για όλες τις δυσκολίες που ε, αντιμετωπίζετε εσείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμιο, οπότε η ισχυρή εποπτεία είναι κάτι απολύτως αναγκαίο. η Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η ΕΣΜΑ και όλοι οι οργανισμοί έχετε πιστεύω κατανοήσει πολύ καλά και πολύ προοδευτικά τα πράγματα μέσω του κανονισμού του ΕΜΙΡ 2.2 και χαίρομαι που θα συνεργαστούμε ελπίζω για το καλό των Ευρωπαίων λαών. Σας ευχαριστώ λοιπόν ξανά και σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα ε, απολαύστε την ημέρα σας στην Washington που θα είναι μεγάλη φαντάζομαι. Εδώ κλείνει το πρωινό κομμάτι της συνεδρίασης της ΕΚΟΝ και θα συνεχίσουμε στις 2 παρατέταρτο.